στη διάταξη. Η Αίγυπτος και κυρίως η υπόθεση του Τζούλιο Ρετζένη. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες καταρχάς. Η κυρία Λόφπιλερ πρώτη. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση των δικαιωμάτων στην Αίγυπτο είναι δραματική και επιδεινώνεται διαρκώς οι Αιγυπτιακές αρχές καταστέλουν θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, στην πραγματικότητα απαγορεύεται η αδίποτε δημόσια διαδήλωση, ασκούνται πιέσεις και απειλές ε, κατά ιδιωτών ή μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οποιοςδήποτε διαφωνεί στην Αίγυπτο κινδυνεύει σοβαρά. Υπάρχουν αυθαίρετες κρατήσεις και προφυλακίσεις χωρίς καμία επαφή με τον ε, έξω κόσμο για εβδομάδες. Το Human Rights Watch έχει καταγράψει πάρα πολλές περιπτώσεις αγνοουμένων κρατουμένων που έχουν, και πολλών που έχουν βρεθεί νεκρύστερα από κράτηση από τις αρχές κράτησης. Δεν είναι φρικτές. Ε, πολλές είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατουμένων που δεν φτάνουν ποτέ ε, μέχρι τα δικαστήρια. Επισκέφθην την ε, Αίγυπτο πριν από μερικές εβδομάδες. Ήταν οι μέρες όπου είχε μόλις ανακαλυφθεί το νεκρό σώμα του ερευνητή Τζούλιο Ρετζένι και ήταν πολλοί μαζί με μένα οι οποίοι καταδίκασαν αυτές, ε, αυτήν και πολλές άλλες ε, παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να φταίνε μέλη του των ε, αρχών ασφαλείας και επιβολής της τάξης για την δολοφονία αυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο για να λειτουργήσει σωστά και το κράτος. Σου δεν υπάρχει αυτό, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ε, μείνουν συνένοχα και να επιτρέψουν αυτή την κατάσταση στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ, Μπέλτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πετρόπη, η δεχθής δολοφονία του κυρίου Ρετζένη θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να δούμε τι προέκυψε από την κοινή έρευνα Αιγύπτου και Ιταλίας. Θα πρέπει να σταθμίσουμε και να μελετήσουμε καλά τα πορίσματα. Έχουν καταστραφεί επίσης πάρα πολλές εκκλησίες και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και την νομοθεσία περί βλασφημίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις για κατάργηση του νόμου περί βλασφημίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει Να δει τι πολιτική ασκεί τελικά απέναντι στην Αίγυπτο. Κοράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Τζούλο Ετζένι ήταν ένας Ευρωπαίος νέος ο οποίος ήθελε να βοηθήσει στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, μιας ελεύθερης κοινωνίας. Η ερευνητική του δουλειά τον οδήγησε σε θέματα που δημιουργούσαν προβλήματα στις Αιγυπτιακές αρχές που ήθελαν να τα αποκρύψουν από την δημόσια σκηνή. Αυτό οδήγησε λοιπόν τον Ρετζένι να βασανιστεί με βάρβαρο τρόπο και να δολοφονηθεί τελικά κάτω από συνθήκες άγνωστες ακόμα. Θα μπορούσε να είναι ο αδελφός μας, θα μπορούσε να είναι ο ανιψιός μας, θα μπορούσε να είναι ο φίλος μας. Παρά τους στενούς δεσμούς που έχουμε με την Αίγυπτο πρέπει να πάρουμε μια αποφασιστική θέση που ε, να ζητά να έχει φως στην ε, δολοφονία του Ρετζένη δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τον ρόλο τον οποίο έπαιξαν οι δημόσιες αρχές. Βλέπουμε τη φωτογραφία του εδώ, την αφιερώνουμε στην οικογένειά του και στους φίλους του. Ζητάμε την αλήθεια για το Ρετζένι. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι θέλουμε την αλήθεια, θέλουμε τη δικαιοσύνη. Έθεσα το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την παρουσία της κυρίας Μογκερίνη η οποία αγνόησε την υπόθεση Ρετζένη. Δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτή. Ε, υπάρχουν ε, όλα σχεδόν οι πολιτικές ομάδες οι οποίες υπογράφουν ε, την συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς έχουμε, θεωρούμε ότι είναι πολύ χαλαρή και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αυτολογοκρινόμεθα. Όταν η Αίγυπτος ήταν υπό την εξουσία του Μόρση και όταν ήταν στην εξουσία οι αδελφοί μουσουλμάνοι, ε, τους έβρισκε η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, προβλήματα στον τομέα της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιου είδους όμως οι αντιλήψεις είναι απαράδεκτες και δυστυχώς ένα καλό άνθρωπο όπως τον νέο αυτό Ιταλό στην ουσία βλέπουμε ότι οδηγήθηκε στην δολοφονία και από θέματα τα οποία ελέγχουν μερικές φορές και αρχές άλλων χωρών. Κύριο Σντεχόφσκι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η υπόθεση του Τζούλιο Ρετζένι πραγματικά πρέπει να θεωρηθεί αποτρόπαια και θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών μας όταν βρίσκονται στην Αίγυπτο. Ε, είναι μια χώρα, η Αίγυπτος, που θεωρούμε ότι είναι στρατικός εταίρος για το μέλλον, που είναι στο πλευρό μας, με την οποία συνεργαζόμαστε. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες υποθέσεις, και σε σχέση και με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταπληξή μας και το σοκ που νιώθουμε. Η Αίγυπτος Όμω, για πρώτη φορά επιτρέπει ε, ομάδα ξένων ερευνητών, Ιταλών στην προκειμένη περίπτωση, και βέβαια σίγουρα είναι ένα καλό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί όμω. Θέλω να καλέσω, καλέσω εκ μέρου του ΕΛΚ τι Αιγυπτικέ Αρχέ να κάνουν πάντα δυνατόν, και το παραλαμβάνω, πάντα δυνατόν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών παραγνώριζοντα εντελώ τι ε, θρησκευτικέ πεπιθήσει, τι πολιτικέ πεπιθήσει. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η περίπτωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Σάκη, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή συνάδελφα, αγαπητέ Επίτροπε, θρυνούμε την απώλεια της ζωής ενός φιέστα του Ιταλού φοιτητή. Όμως ε, η βασανισμή είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο και γι' αυτό θα πρέπει να ασκήσουμε έντονες πιέσεις ε, για την αποδόση δικαιοσύνη, αλλά και για όλες τις άλλες ε, υποθέσεις. 1.700 περιπτώσεις με βάση ΜΚΟ ε, κατά την προηγούμενη χρονιά. Είναι σαφές ότι οι αρχές επιβολής του νόμου προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας Ιταλών Αιγυπτίων, αλλά να είναι αποτελέσματα αποτελέσματα μια αξιόπιστη έρευνα κάτι που δεν συμβαίνει πάντα στην Αίγυπτο και βλέπουμε ότι λιγότερο επιβάλλεται δικαιοσύνη, περισσότερο υπάρχει ατιμορρησία. Με ανησυχεί επίση ε, η κυβέρνηση Ασίζη και η προπαγάνδα τη ε, που στρέφεται επίση κατά των αντιφρόντων, κατά των πολιτικών αντιπάλων. Το 2013 πάνω από 22.000 άνθρωποι ε, μπήκαν φυλακοί με βάση τι ίδιε Αιγυπτιακέ αρχέ. Καιρό πια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσει το αναστημά τη να ακουστεί η φωνή της και τουλάχιστον ε, να μην ε, επιτρέψει η διευκολύνη ακόμη περισσότερο της ε, παραβίασης των δικαιωμάτων με τα προγράμματα ανταλής. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, οι αρχές των Αιγυπτίων και διερωτώ με ειλικρινά τα διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν γιατί δεν διαπνέουν και δεν καθοδηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι για το 2011 τα γεγονότα και τα δάγματα θα πρέπει ακόμα να σκαθοδηγούν. Ευχαριστώ. Πέρασαν πέντε εβδομάδες από το θάνατο του Ρετζένη και κάθε εβδομάδα οι πτιακές αρχές αλλάζουν την ιστορία τους γιατί από ό,τι φαίνεται πρόκειται για μια πολιτική δολοφονία μετά από διαταγή του ε, καθεστώτος Αλσίση. Η κυβέρνησή μου δυστυχώς δεν βρήκε την αξιοπρέπεια να καταγγείλει αυτή την κοροϊδία και να πάλι τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται διακόπτοντας τις οικονομικές σχέσεις με το καθεστώς ε, του Αλσίζη στο όνομα υποτίθεται της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ένα δικτάτορα ο οποίος έχει σαν βασικό μέσο διακυβέρνηση την καθημερινή τρομοκρατία. Σήμερα το Κοινοβούλιο κάνει το αξιοπρεπές κάτι πεπές αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει εμείς να καθεστώτα όπως του Αλσίση και του Ερντογάν να τα καταγγέλουμε. Και δεν πρέπει να τους δίνουμε πόρους για να καταπιέζουν τους λαούς τους. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο καταδικάζει τον βασανισμό και τον θάνατο του Βεντζένη, αλλά ζητά να δοθούν στις Ιταλικές αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να υπάρξει μια διαφανής αντικειμενική ανακριτική διαδικασία. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική της εξαφάνισης των αντιφρονούντων μετά από βασανιστήρια. Η Αίγυπτος θα πρέπει επίσης να απελευθερώσει τους κρατούμενους για λόγους ελευθερίας έκφρασης, να επιτρέψει την λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών και των ελεύθερων συνδικάτων. Στρέφομαι προς εσάς κύριε Χάν. Λέγω ότι η Αίγυπτος πράγματι είναι ένα σημαντικό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το τίμημα πρέπει να είναι ελεγχόμενο δεν θα κλείσουμε τα μάτια λοιπόν σε αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ, αλλά φοβάμαι ότι ε, ε, έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο στη διάθεσή μας. Ακούσαμε τους εισηγητές, ακούσαμε τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων και θα πάμε τώρα στον συνάδελφο κύριο Πόλτσακ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει φοβερές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί η αδίποτε δικαιολογία για τις παραβιάσεις από πλευράς των εκπροσώπων των αρχών των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η περίπτωση του Ρετζένη είναι ε, τραγική. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια θεσμοθετημένη πρακτική να ξεφορτώνονται οι κρατικές αρχές οποιονδήποτε τις ενοχλεί. Οποιονδήποτε δεν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που έχουν ορίσει για μια χώρα σύγχρονη, όπως θέλει να είναι η Αίγυπτος, αν κρίνουμε από το Σύνταγμα του 2014 που ενέκρινε. Δεν είναι όμως σύγχρονη χώρα και οι λόγοι είναι προφανείς είναι οι αντιφάσεις μεταξύ του γράμματος και της εφαρμογής του συντάγματος. Κατοντάδες χιλιάδες ε, χιλιάδων ανθρώπων έχουν εξαφανιστεί στα χέρια των αρχών, πολλές φορές βρεθεί δολοφονημένοι. Είναι προφανές ότι δεν πληρεί τα βασικά κριτήρια για ένα δημοκρατικό καθεστώς η Αίγυπτος. Ευχαριστώ. Δημοκράτες, κύριε Ντεμόντε. Μιλάμε για ένα ψήφισμα το οποίο αφορά στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα όμως ασχολούμαστε με την υπόθεση του θανάτου του Τζούλο Ρετζένη, ένας συμπατριώτης μου ε, ερευνητής ε, με όλο το μέλλον δικό του, είχε πάει στο Κάιρο για να εμβαθύνει τις μελέτες του, αλλά δυστυχώς μετά από απερίγραπτα βασανιστήρια έχασε την ίδια του τη ζωή. Το Κάιρο η κυβέρνηση μας έδωσε πίσω ε, το ίδιο το σώμα του Ρετζένη αλλά δεν μας έδωσε τα στοιχεία της αλήθειας που απαιτούνται. Νομίζω ότι οφείλουμε σε αυτόν, στην οικογένειά του, στους φίλους του, και στην κοινότητα του Φιουμιτσέλο από όπου προέρχεται να πούμε την αλήθεια και ιδιαίτερα το οφείλουμε σε όλους τους νέους που πιστεύουν στην δημοκρατία, στο δικαίωμα στη ζωή το οποία κανένας δεν μπορεί να σταματήσει. Ο κύριος Μπούχνερ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα οι αρχές του κράτους δικαίου είναι κεντρικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει, έχουν τη θέση τους και στη στρατηγική για το εμπόριο. Πρέπει δηλαδή τις αξίες αυτές να τις στηρούν και οι εμπορικοί μας εταίροι, οι χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε συναλλαγές. Ωστόσο, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή παραβιάζονται, σε όλες τις χώρες δηλαδή. Ιδιαίτερα όμως για την Αίγυπτο πρέπει να πούμε ότι έχει ε, τραγικά επιδεινωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο πως θέλει να απαγορεύσει αδίποτε δημόσια εκδήλωση απόψεως, ακόμη και διαδηλώσεις οι οποίες θα υποστήριζαν την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα το οποίο έχουμε να εγκρίνουμε σήμερα έρχεται την κατάλληλη στιγμή και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντως να δώσει έμφαση στην ε, τήρηση των όρων που συμπεριλαμβάνουμε στις εμπορικές μας συναλλαγές με την Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ. Ήρθαμε εδώ για να καταδικάσουμε μία βαρβαρότητα, μία παράδεκτη δολοφονία. Είναι απαράδεκτοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι Αιγυπτιακές αρχές για να μην πουν την αλήθεια από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Δεν αρκεί να ζητήσουμε η κυβέρνηση αυτή να ρίξει φως. Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως ε, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο. Ε, ο ακραίος, ε, η ακραία τρομοκρατία δεν θα πολεμηθεί μέσω της κρατικής τρομοκρατίας. Σήμερα λοιπόν συνάδελφοι δεν χρειάζεται να κάνουμε το μνημόσυνο του Τζούλιο, θα πρέπει να δράσουμε και ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Θέλουμε αλήθεια και δικαιοσύνη για τον Τζούλιο Ρετζένη. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λόπεθ για ένα λεπτό. Εδώ είμαστε για να καταδικάσουμε το χαμό του Τζούλου αλλά και για να θυμίσουμε πώς πέθανε όπως πολλοί ε, άλλοι ε, ακτιβιστές στην Αίγυπτο ε, πριν από πέντε χρόνια και στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Είμαστε δύο να πούμε επίσης ότι στο μέλλον οι διεθνείς σχέσεις και ο σεβασμό στα θύματα συνεπάγονται την αποκάλυψη της αλήθειας ε, που ε, στην περίπτωση αυτή συγκαλύπτεται. Δεν είναι απομονωμένο το περιστατικό, είναι μακρός ο κατάλογος δικηγόρων, ακτιβιστών, υπερσπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων οι οποίοι ε, μπήκαν στη φυλακή και πολλοί βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν στην Αιγυπτό τα τελευταία χρόνια. Είμαστε εδώ για να πούμε σήμερα ότι δεν πήγε μάταιος αυτός ο θάνατο ότι θα μας εμπνεύσει ο χαμός αυτού του νέου κατά τρόπον ώστε σήμερα να πούμε ότι δεν ε, θα κλείσουμε πια τα ε, μάτια μας απέναντι στην αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Είναι στρατηγική, όχι σχέση μας με την Αίγυπτο, αλλά η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε στις αρχές. Αιγύπτο, ευχαριστώ. Κύριος Καν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταδικάζω απερίφραστα την ε, αποτρόπαιη δολοφονία του Τζούλιου Ρετζένη και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους οικείους του. Πρέπει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, η οποία αποτελεί συνέχεια μια σειρά εκατοντάδων μυστηριωδών εξαφανίσεων από την ανάληψη τη εξουσία του στρατού ε, στην Αίγυπτο. Είναι πολύ όχι μόνο οι Αλοδαποί, αλλά και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και δεν έχουν κληθεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη εκπρόσωποι των αρχών που έχουν ασκήσει υπερβολική βία και οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο και σε θανάτωση πολιτών. Ε, πρέπει λοιπόν να ανατραπεί αυτή η νομοθεσία η οποία οδηγεί σε μια εσωτερική καταστολή. Πρέπει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση να πιστεί να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι και τώρα. Ύστερα από το σύντομο αυτό κατάλογο παρεμβάσεων θα περάσουμε σε ένα μακροσκελέστερο κατά πολύ κατάλογο ε, συναδέλφων που έχουν στήσει το λόγο, που δυστυχώ όμω δεν μπορώ να εικονοποιήσω του πάντε για λόγου χρόνου. Κύριο Σταγιάννη έχει το λόγο. Η Αίγυπτος είναι βασικός συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική χώρα για τη σταθερότητα στην Μεσογειακή Λεκάνη. Όμως δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τις μας να υπονομευθούν για λόγους εμπορικούς ή για λόγους πολιτικούς. Ο διάλογος με μια χώρα σαν την Αίγυπτο βασίζεται και στην απαραίτητη ε, συνεργασία ε, και στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εκτών των συνόρων της. Ε, απαιτείται περισσότερη δράση ε, και ε, από την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική δράση. Θα θέλαμε να τη δούμε πιο δραστήρια και στην, στους δύο Ιταλούς πεζοναύτες οι οποίοι κρατούνται στην Ινδία ή στην περίπτωση των δύο Ιταλών εργαζομένων που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεχθήκατε και τα χειροκροτήματα των συναδέλφων. και ως Καπούτο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει έτσι ώστε να αρχιθεί φως στον τραγικό θάνατο του Ρετζένη. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, δεν υπάρχει βολική αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη στον Ρετζένη θα πρέπει να γίνει γνωστό θα πρέπει η Ευρώπη να ζητηθεί να μάθουμε επιτέλους τι συνέβη στον Ρετζένη και τι γίνεται με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Είναι σημαντικός εταίρος της Ένωσης η Αίγυπτος, αλλά πρέπει να σέβεται ε, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία ε, της πίστης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το οφείλουμε στον Ρετζένη, το οφείλουμε στην αξιοπρέπειά μας. Ο κύριος Μαριάς. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Η δολοφονία στην Αίγυπτο του Τζούλιο Ρετζένι, ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεχύλισε το ποτήρι. Καταδικάζουμε τη δολοφονία του Τζούλιο Ρετζένι. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους φίλους Ιταλούς συναδέλφους που πήραν πριν λίγο το λόγο. θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα στην αίγυπτο η οποία οφείλει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να αντιληφθεί η αιγυπτιακή ηγεσία ότι η καταπίεση των δημοκρατικών ελευθεριών και του αιγυπτιακού λαού αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των τζιχαντιστών οι οποίοι καραδοκούν για να πάρουν τη ρεβάνς είναι δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να εκφράσει την καταδίκη της για τη δολοφονία του τζούλιο ρετζένι. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, εκφράζω και εγώ τη βαθύτατη οδύνη μου προς τους οικείους του Ρετζινη και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη και άνευ προϋποθέσεων έρευνα του θανάτου του. Αλλά είναι μία μόνο αυτή η περίπτωση από τις εκατοντάδες χιλιάδων περιπτώσεων και δεν θέλω να καταλαβώ καλύτερα τι κάνουν οι αρχές στην Αίγυπτο. Και χτες ακόμη έγινε λόγος για την εταιρική σχέση με την Τουρκία και τα όσα πράττει ο Ερντογάν όπου θα σπεύσουμε να το απελευθερώσουμε τη θεώρηση του διαβατηρίου και να το ανοίξουμε κεφάλαια. Το ίδιο με το Καζακστάν, όταν ξέρουμε με τι κατασταλτικό καθεστώς έχουμε να κάνουμε. Και τώρα έχουμε και την Αίγυπτο. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικός εταίρος. Αλλά επιτέλους κύριε Επίτροπε, δώστε μας κάποιους ε, οδηγούς, κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μας με την Αίγυπτο στο μέλλον για να έχουμε μια καλή και ισχυρή εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Κούζο. Ευχαριστώ. Πριν 10 χρόνια οι συνδικαλίστες από τη Μαχάλα μας ε, έδειξαν ε, ότι στην Αίγυπτο ζητείται δικαιοσύνη, ψωμί, ο Μουμπάρακ, ε, κακομαθημένος από τα τη μέλη της Ευρώπης και της ΕΠΑ. Δυστυχώς ούτε δικαιοσύνη, ούτε ψωμί, ούτε ελευθερία έφτασε στη χώρα, αλλά άλλο πραξικόπημα. Πάνω από 100 δις πληρώνει η Αίγυπτος στο στρατό και στον οποίο πουλάνε όπλα οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το καθιστό έχει πάνω από 1.700 καταδίκες και έχει ε, εκτελέσει ε, εκατοντάδες ανθρώπους. Ε, ο, Τζουλιάνο, ο Τζούλιο Ρετζένι, ο οποίος βασανίστηκε φρικτά, δολοφονήθηκε όλα, αυτά σε μια χώρα στρατηγικό εταίρο της Ένωσης. Δεν μπορεί να το αφήσουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό μπορεί όμως να συμβεί και το φοβάμαι πολύ. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το κάνει πάντα όταν τη συμφέρει και μόνο. Ευχαριστώ. Δεν Και τώρα ο κύριος Μπονάνο, παρακαλώ. Sì, signor Presidente, io... την περίπτωση, σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση, θα ήθελα να πω... Θα ήθελα να πω ότι αν πράγματι η Ευρώπη θέλει να είναι ενωμένη, πρέπει να πει στην Αίγυπτο ή θα μας πει την αλήθεια για αυτό που συνέβη στο Ρετζένι ή αλλιώς θα μπλοκάρουμε κάθε σχέση οικονομική και διπλωματική. Αυτό θα αρκέσει έτσι ώστε να καταλάβει η Αίγυπτος ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει την οικογένεια του Ρετζένι, τον ίδιο τον Ρετζένι που δεν είναι πια ανάμεσά μας και να μην συνεχίσει να δίδει τέτοιες απαράδεκτες ε, απαντήσεις ε, κάθε φορά αντίθετες η μία με την άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι εδώ διακυβεύεται η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία της Ευρώπης πρέπει εμείς να εμβαθύνουμε την έρευνα, μια έρευνα η οποία είναι ελεγχόμενη, μια έρευνα η οποία δυστυχώς δεν την χάνει των απαραίτητων εγγύσεων. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια ε, στην δολοφονία του Τζούλιο Ρετζένι. Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος έψαχνε, ε, ερευνούσε ένα σύστημα για να καταλάβει την λειτουργία του θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προσπάθειες ε, από την κυρία Μογκερίνη για να ε, μάθουμε την αλήθεια και γιατί όχι να διακόψουμε στην παρούσα φάση τις εμπορικές σχέσεις γιατί η αναζήτηση της αλήθειας είναι προτεραιότητα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Χάουιτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως Βρετανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου εκφράζω την ε, συμπάθειά μου και τα συλληπιτήριά μου στους Ιταλούς συναδέλφους αλλά και την οικογένεια του Τζάνι Τζούλιο Ρετζένι. καλώς και όλων αυτών που έχουν πέσει θύματα αντίστοιχης βίας στην Αίγυπτο. Θα παρακαλέσω τον Επίτροπο να με ρημνήσει ιδιαίτερα για τις εξαγωγές, για τη ρύθμιση των εξαγωγών εξοπλισμού παρακολουθήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις και σε επίπεδο Γερμανίας και σε επίπεδο της ομάδας των hackers που, είναι, ε, που εδρεύει στην Ιταλία. Πληροφορίες λοιπόν οι οποίες συλλέγονται και με πολύ ε, υψηλά κονδύλια για τις παρακολουθήσεις αναπτύσσει και η Αίγυπτος χωρίς καμία επαλήθευση από ανεξάρτητη αρχή ή το κοινό. Παραβαίνουν βέβαια τις αρχές των ΗΕ και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων τέτοιες ε, δράσεις και δεν πρέπει σε αυτό να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Giulio Regeni tragikus és brutális halálának körülményeit független és Ήταν βίαιος ο θάνατο ε, του Τζούλο Ρετζένη και αυτό θα πρέπει να το ερευνήσει μια αμερόληπτη ε, ερευνητική ομάδα. Φοβάμαι βέβαια ε, ότι δεν πρόκειται να χυθεί άπλητο φως αυτήν την υπόθεση ποτέ. Ο νεαρός αυτό σίγουρα δεν έπεσε θύμα ενός εγκληματο του κοινού ποινικού δικαίου. Αλλά αυτό ο θάνατο οφείλεται στις πολιτικέ του απόψει και στην δράση του και αυτό είναι απαράδεκτο. Και ακόμη και αν έγινε σε αυτή τη χώρα. Ε, Ιδίω όταν βλέπουμε ότι πέντε χρόνια μετά την Επανάσταση ε, είναι ακόμα ε, σκοτεινά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, ίσως ακόμα πιο σκοτεινά και θολά. Η υπόθεση αυτή πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ. E Αλήθεια και δικαιοσύνη για τον Ρεντζένι είναι το καθήκον όλων μας, αυτό πρέπει να επιδιώξουν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι καμία οικονομική πραγματικότητα δεν θα συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες παρακολούθησης, καταστολής βασανιστήριων σε μια χώρα σαν την Αίγυπτο επανειλημμένα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το υπενθυμίζει αυτό το κοινό μας ψηφίσμα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε με την κατάσταση αυτή με όλες μας τις δυνάμεις. Νομίζω ότι η περίπτωση του Ρετζένη θα πρέπει να μας οδηγήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει ιδιαίτερα για τους νέους που συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα και θέλουν να αλλάξει ο κόσμος. Ο Τζούλιο με τις έρευνές του ε, πλήρωσε με τη ζωή του μάλλον την έρευνα αυτή, την αναζήτηση της αλήθειας. Ugyanúgy vélekedett ebbe a kérdésben. Öné a viszont lehetősége parancsoljon. Φαντάζομαι ότι όλοι ε, ότι έχουν την ίδια άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Θα σας δώσω τώρα σε εσά ε, το λόγο, πίτρο, πως Ναι, πραγματικά ε, είναι κοινή η άποψη μεταξύ όλων. Όλους μας ε, σώκαρε η ανακάλυψη της ορού του Τζούλιο Ρετζένι στο Κάιρο. Είχε εξαφανιστεί από τον Ιανουάριο, βρέθηκε νεκρός αρχές Φεβρουαρίου. Ήταν ένας νεαρός φοιτητής στο Κάιρο. Αυτή, αυτός ο χαμός είναι μια προσωπική απώλεια τραγωδία για όσους τον γνώριζαν, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα θεσμικά όργανα και για τον απλό κόσμο. Νομίζω το είπαν όλοι οι σημερινοί Η κυρία Μογκερίνη δύο φορές ε, έθεσε το ζήτημα της δολοφονίας Ριτζένη ε, στην κυβέρνηση του ΣΥΣΥ και ζήτησε να γίνει μια ανεξάρτητη ε, διαφανής έρευνα σε στενή συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές ώστε να χυθιάπλε το φως ε, στις ε, συνθήκες του θανάτου του και για την προσαγωγή των ε, θητών, των ενόχων στην δικαιοσύνη. Υπήρξαν θημερεί επαφές με τι Αιγυπτιακέ αρχέ και το Φεβρουάριο. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και η ΕΙΕΔ παρακολουθούν την υπόθεση στενή συνεργασία και συνεννόηση με την Ιταλική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και ε, πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα, ε, συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου. Να σας δώσω και ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα. Ε, είχαμε διάφορες προσπάθειες για το κλείσιμο του κέντρου Ναντίν, το οποίο παρέχει θεραπευτική υποστήριξη σε θύματα βασανισμών η προστασία ε, δημοκρατίας, ε, ε, η ελευθερία, το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδης λύθη των πολιτικών στο 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση επανέν ξεκίνησε τις διμερείς σχέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης η οποία ήταν σε αναστολή από το 2010 και αυτός το κάναμε γιατί θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στον τομέα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και να έχουμε συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος πέρυσι τον Νοέμβριο στο Κάιρο ξεκίνησε επίσης ο διάλογος για θέματα ε, πολιτικά και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από πέντε χρόνια. Υπάρχουν στενές επαφές και με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και τις οργανώσεις και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Μογκερίνη ζήτησε πριν από τέσσερι μήνε ε, να επισκεφθεί αυτέ τι οργανώσει ε, στο Κάιρο. Επίση, με τα κράτη-μέλη εξεργαζόμαστε μία δήλωση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Αιγυπτό, την οποία θα εκφωνήσουμε στι 15 Μαρτίου στη Γενέβη. Οπότε και συνεδριάζει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ε, Ο ειδικό απεσταλμένο των δικαιωμάτων θα επισκεφθεί τη χώρα του επόμενου μήνε, ώστε να υπάρξει συνεχής, συνεχιζόμενη συνεργασία με την Αίγυπτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από κοινού και με τις ταλικές αρχές, ώστε να βγει στο φως η πλήρης αλήθεια και οι δράστες για, οι υπεύθυνοι για, για το ε, απάνθρωπο βασανιστήριο και το θάνατο του Ρετζέν να προσαχθούν ενώπιν της δικαιοσύνη. Επίσης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τέτοιες απαράδεκτες τραγωδίες στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ζητούμε ε, και να ε, επιμένουμε για την η πλήρη εφαρμογή των, των, του συντάγματο του 2014 μεταρρυθμίσει στον τομέα ε, τη διακυβέρνηση του κράτου δικαίου. Θέλουμε πρόοδο στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί αυτά είναι ε, προσδοκίες του ίδιου του λαού ε, της Αιγύπτου για τη σταθερότητα και για την ευημερία, την ειρήνη. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ε, στο πλαίσιο της συνεργασία μας συνεργαζόμαστε και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και τις οργανώσεις κοινωνία των πολιτών για την αντιμετώπιση ιδίω όλων αυτών των ζητημάτων και για, την, για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτός είναι και ο στόχος μας ε, γενικότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Έχουμε 8 ψηφίσματα.